Ε, chers amis, est-ce que vous savez que vous pouvez utiliser les... Ε, υπάρχει και διερμηνία στη διάθεσή σας, ενημερώνει Πρόεδρος. Merci beaucoup. dear colleagues, I would like... Αγαπητοί συνάδελφοι, να καλωσορίσω τους ε, προσώπους των συλλόγων του Κλίσι Σούμπουα που θέλουν να μοιραστούν μαζί μας κάποιες εντυπώσεις για την κατάσταση στις αστικές περιοχές κοντά στο Παρίσι. Όπως ξέρετε, μία αντιπροσωπεία της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης επισκέφθηκε τη Γαλλία και ο στόχος ήταν ε, να εξεταστεί η εφαρμογή της πολιτικής συνοχής σε κάποιες γαλλικές πόλεις και να δουν συγκεκριμένα παραδείγματα παρέμβασης της πολιτικής συνοχής σε τοπικές αστικές κοινότητες. Δεν είχαμε χρόνο εμείς να μεταβούμε στο κλεισί Σουμπουά, έτσι λοιπόν θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο να σας ακούσουμε για να κατανοήσουμε καλύτερα και πώς αντιλαμβάνεστε εσείς την κατάσταση σε αυτές ε, τις ε, μη ευνοημένες περιοχές και όπως ξέρετε τώρα προετοιμάζεται η μελλοντική πολιτική συνοχής ε, και η αστική ανάπτυξη είναι πολύ ψηλά στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της περιφερειακής πολιτικής και γι' αυτό θεωρούμε ότι και επίσκεψή σας εδώ αποτελεί ευκαιρία να λάβουμε υπόψη και τη δική σας ε, δουλειά και τις ανησυχίες που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Ε, δεν ξέρω αν η κυρία Καρμαντέλη θέλει το λόγο και κατόπιν θα ακούσουμε και εσάς. Πρόεδρε. Αυτοί οι νέοι και οι λιγότερο νέοι ε, που προέρχονται από το κλειστή Σουμπουά έκαναν μία έκκληση με ισχυρές ε, διεκδικήσεις και αυτή την έκκληση την απευθύναν στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Μπαρός, ο οποίος τους είπε ότι λόγω έλλειψης χρόνου δεν μπορούσαν να τους δεκτεί και εγώ σας ευχαριστώ πρόεδρε που εδώ αφιερώνετε το χρόνο και που απαντήσατε θετικά στην έκκλησή τους και χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκονται ενώπιόν μας εδώ σήμερα προκειμένου να μας εκφράσουν τα προβλήματα και τις ανησυχίες τους και θα ήθελα να σας καλωσορίσω. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο κύριε Σίσα. Μικρόφωνο παρακαλώ. Bonjour, déjà merci de nous, euh, nous Σας ευχαριστώ για την υποδοχή σας εδώ. Εμεί ε, απευθύναμε μια έκκληση στον κύριο Μπαρόσο που δημοσιεύτηκε στη Λιμπερασιόν ε, στις 27 ε, Οκτωβρίου και θα σας τη διαβάσω έτσι λοιπόν μια έκκληση των κατοίκων του Κλεισί στο Ζωζέ Μανουέλ Παραντουράου Μπαρόσο. Εμείς θεωρούμε ότι δεν ισχύει πλέον η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, η στρατιωτική, αλλά ε, ισχύει η κοινωνική κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και έτσι λοιπόν υποχρεούμαστε να πούμε σε όλους ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει. Το κράτος είχε δεσμευτεί να ε, θέσει σε εφαρμογή ένα πραγματικό σχέδιο Μάρσαλ, ε, ενεργοποιώντα όλα τα Υπουργεία έτσι ώστε να ισχύει το δίκαιο σε εμά όπου και παντό εμεί σήμερα πολιτιστική, αθλητική και οργάνωση των πολιτών ε, του Εκκλησίου Μπουάθ ε, βλέπουμε ότι ε, δεν ισχύουν υποσχέσεις που μας είχαν δώσει οι θύνοντες της χώρας και με την καθημερινή διαχείριση της κοινωνικής μισέργειας εμείς, εμείς προσπαθούμε να εμποδίσουμε μία μεγαλύτερη έκρηξη θέλουμε να πούμε όχι στη βία αλλά να συνεχίσει το κράτος να μας λέει όχι τότε πάντοτε η βία θα έχει την τελευταία λέξη. Υπάρχει μία άλλη φωνή, πιο δημοκρατική και πιο δίκαιη, του σεβασμού και της αναγνώρισης. Γνωρίζετε τις προσπάθειες των κατοίκων της συνοικίας μας που αποτελούν τμήμα της γαλλικής κοινωνίας ε, και ε, καθημερινά βλέπουμε να υπάρχει η δημιουργία των γκέτο, οι δεσμεύσεις και υποσχέσεις που δόθηκαν μετά τι τις αντιπαραθέσεις και την τραγωδία ε, έχουν να κάνουν με τις μελλοντικέ ε, γενιές που θα είναι ο λαός ε, της δημοκρατίας. Δεν μπορούμε να θυσιάσουμε όλα αυτά στο βωμό ε, του εγωισμού μας ξεχνά ε, η χώρα μας και γι' αυτό εμείς απευθυνόμαστε στην Ευρώπη για να αναλάβει τις ευθύνες της και να δείξει σεβασμό στους ανθρώπους και στους λαούς και ε, με αυτή την αλληλέγγυα, ε, σε αυτή την αλληλέγγυα Ευρώπη απευθυνόμαστε και ζητάμε από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μας δεκτεί για να, μπορούμε, να, να μπορέσουμε να τους εκθέσουμε τα σχέδιά μας και ζητούμε επίσης και από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κυρίως της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης να δεχτούν την επίσκεψή μας. Ε, η εξέγερση του 2005 είχε ε, ε, την κατάληξη τουλάχιστον τα άτομα που σήμερα θα ήταν 22 και 25 χρονών να μην χαθεί η φωνή τους σήμερα. Δεν θα χανόταν. Θα δώσω το λόγο στο συνάδελφο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριε Ευρωβουλευτέ. Από το 2005 δεν έχει αλλάξει τίποτα στο προάστιό μας. Υπάρχει μια ε, όλο ένα και μεγαλύτερη αύξηση του συγκετοποίησης. Υπάρχει μια αναδιάρθρωση της ε, φτώχειας και των κοινωνικών και ταφικών ανισοτήτων. Σε αυτή τη γειτονιά λοιπόν ε, δεν έχουμε καταφέρει να θέσουμε ένα τέλος στην επικινδυνότητα και έχει ε, πια γίνει ο φαταλισμός ε, μέσα στα πλαίσια και της οικονομικής και κοινωνικής ε, κρίσης σε μια πραγματικότητα που συνεχώς επιδεινώνεται. Με βάση όλα αυτά λοιπόν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι ενώσεις και οι τοπικές και οι τοπικοί φορείς είναι αδύναμοι μπροστά στο κράτος. Δεν έρχονται σε εμά ε, οι χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχουν άμεσες επιπτώσεις για την εκπαίδευση των νέων στη γειτονιά αυτή. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν αυτή τη δύσκολη κατάσταση και την κοινωνική και οικονομική κρίση, θέλουμε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο Marshall για τα προάστια των μεγάλων αστικών ε, περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να υπάρχει ένα νόημα στη δράση μας αλλά και να δοθεί νέος ε, ρυθμός στην ευρωπαϊκή πολιτική. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένη δουλειά ώστε να ενσωματώσουμε τους ε, ανθρώπους αυτούς στην κοινωνία μας, να δώσουμε ε, στους κατοίκους των προαστίων αυτών τη δυνατότητα να αλλάξουν την καθημερινή τους ζωή, να έχουν ένα μέλλον για τα παιδιά τους. Θεωρούμε λοιπόν ότι η κατασκευή ε, κάποιων ε, κατοικιών θα μπορούσε να μειώσει τις δυσκολίες ε, όπως επίσης και οι καλύτερες μεταφορές έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος για θέσεις απασχόλησης, πανεπιστήμια και μέρη όπου η κοινωνική ζωή λαμβάνει χώρα. Όλα αυτά τα στοιχεία μας ανησυχούν γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα για τη χώρα μας, ε, τη Γαλλία. Ποια είναι τα στοιχεία που θα πρέπει και τα εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε ε, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τη Γαλλία και να τη βοηθήσουν και όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούμε ότι η κατάσταση είναι πραγματική και θέλουμε μια συνεργασία επικοδομητική. Ίσως θα μπορούσε να μας βοηθήσει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όμως δυστυχώ δυστυχώς ε, η δυσκολία στην οποία βρισκόμαστε είναι κάτι το οποίο δεν επιλύεται. Πρέπει λοιπόν εμείς να παίξουμε το ρόλο που χρειάζεται να παίξει το κράτος, όπου αυτό δεν είναι παρόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ε, ο κύριος Σαμίρα Μπάς θέλει να λάβει το λόγο. Καλημέρα σας ε, κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές. Είμαι στον εκπαιδευτικό κόσμο. Είμαι ε, καθηγητής και ε, δάσκαλος. Συγκεκριμένα δουλεύω με παιδιά 6, ε, παιδιά 6 έως 10 ετών και τώρα δουλεύω και με μαθητές 16 έως 20 ετών. Μέσα από αυτήν την εμπειρία συνειδητοποίησα τα εξής. Η ποιότητα της διδασκαλίας στη Γαλλία μειώνεται και κύρια στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ε, κοινωνική ανάπτυξη του κάθε ατόμου χάνονται. Γι' αυτό το λόγο ένα μεγάλο μέρος αυτών των μαθητών, ε, αυτών των ε, νέων φεύγουν από το σχολείο χωρίς πτυχίο στα 16 τους χρόνια με συνθήκες επισφάλειας. Δεν έχουν προσόντα, δεν μπορούν να, να χρησιμοποιήσουν αυτά που ξέρουν στην αγορά εργασίας και δεν μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Αυτό προέρχεται από πολλούς παράγοντες. Η έλλειψη κυρίων ε, στοιχείων, θεμελιωδών στοιχείων, όπως η ανάγνωση, η γραφή, η αριθμητική. Δεν υπάρχουν δράσεις που να στρέφονται προς τα πολιτιστικά ε, από τη νεαρή ηλικία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά και οι νέοι να μην μπορούν να διαβάσουν σωστά και να μην μπορούν να εκφραστούν σωστά. Και αυτό εξηγεί και το χαμηλό επίπεδο ε, επιτυχίας των ατόμων που μένουν στις πιο επομβαθμισμένες ε, ε, περιοχές. Αυτό είναι πολύ δύσκολο και αντιπροσωπεύει 150.000 παιδιά που φεύγουν από το κόσμο του σχολείου αυτοί οι νέοι βρίσκονται σε συνθήκες ανεργίας χωρίς να έχουν ξεκινήσει καν να εργάζονται ή καταλήγουν σε επισφαλείς θέσεις εργασίας. Αυτό οδηγεί τους νέους αυτούς σε συνθήκες αποκλεισμού, κοινωνικού, ε, γεωγραφικού ή και οικονομικού αποκλεισμού. Είναι σημαντικό να δούμε το εκπαιδευτικό σύστημα από τη βάση του. Πρέπει να ε, ενισχυθούν τα κύρια χαρακτηριστικά, τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του σχολείου. Πρέπει να προσαρμοστεί το εκπαιδευτικό σύστημα στην αγορά ε, εργασίας. Πρέπει να ενισχυθούν οι κλάδοι που ε, δημιουργούν θέσεις εργασίας, όπως θέσεις εργασίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, όταν οι μαθητές φεύγουν από το σχολείο στα 16 τους χρόνια χωρίς να μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους επειδή δεν έχουν πτυχίο ή επειδή δεν υπάρχει διαθέσιμη θέση ε, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα όπου θα μπορούσαν να ακολουθήσουν τον κλάδο ε, που θέλουν, πρέπει να απευθυνθούμε στην κοινωνία έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η προοπτική του μέλλοντος γιατί το, οι νέοι δεν βρίσκονται τότε μόνο σε επισφαλείς συνθήκες, αλλά και σε συνθήκες αποκλεισμού. Πρέπει να δούμε ποια είναι τα επαγγέλματα που χάνονται και να ε, επενδύσουμε στις νέες τεχνολογίες, στα πράσινα επαγγέλματα και στα επαγγέλματα που έχουν μέλλον στην Ευρώπη, έτσι ώστε να δημιουργηθούν και αντίστοιχοι ε, κλάδοι στην εκπαίδευση γιατί προς το παρόν αυτοί οι κλάδοι δεν υπάρχουν ε, στις αγροτικές περιοχές και στις πιο απομακρυσμένες περιφέρειες. Η συνεχιζόμενη κατάρτιση τώρα. Πολλά άτομα μέσα από την επαγγελματική τους πορεία αποφασίζουν να αλλάξουν ε, επάγγελμα στα 40 τους χρόνια, για παράδειγμα αυτοί οι άνθρωποι, για παράδειγμα, δεν γνωρίζουν τις νέες τεχνολογίες, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν υπολογιστή, δεν μπορούν να γράψουν ένα mail. Αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε οικονομική ανεργία και δεν μπορούν να ε, ε κατευθυνθούν σε νέες καριέρες, νέα επαγγέλματα, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες Και επίσης πρέπει όλα τα μέτρα να απευθύνονται σε όλες τις ηλικίε. Γιατί όλες οι ηλικίε αφορούν μια ε, γενιά που βρίσκεται σε κίνδυνο. Η οποία ζει και επιβιώνει χάρη στις άλλες γενιές. Και τέλος θα ήθελα να πω ότι όλα αυτά δεν είναι δύσκολο να εφαρμοστούν. Πρέπει όμως να υπάρχει μια γενική ε, πολιτική σε όλη την επικράτεια έτσι ώστε να μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτά τα ε, μέτρα με ενεργό τρόπο και να μην χανόμαστε μέσα στη γραφειοκρατία. Ευχαριστώ. Ε, Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να προσθέσει κάτι. Ναι, επανέλθω στην ημερήσια διάταξη τα θέματα της αστικοποίησης και της ε, στέγασης. Σας ζητάμε να μην κάνετε το λάθος που έκανε η Γαλλία στη δεκαετία του 60, 60 που θεωρούσε ότι η στέγαση και η αστικοποίηση είναι θέμα κατοίκων και περιβάλλοντος. Ε, πριν από αυτό υπάρχουν λοιπόν πριν από το θέμα της στέγασης ε, θα πρέπει να δούμε τον ανθρώπινο παράγοντα ε, έτσι ώστε να έχουμε την ανθρώπινη διάσταση που θα μας καθοδηγεί στο θέμα της αστικοποίησης και της στέγασης. Η ανθρώπινη διάσταση, ο άνθρωπος στο κέντρο του, του ζητήματος της αστικοποίησης που ζει σε μία πόλη, σε μία ε, συνοικία, δεν είναι αυτός που απλώς κατοικεί, ε, ζει σε αυτή, θέλει να, να διασκεδάσει, να, να χρησιμοποιήσει τις μεταφορές, να κάνει ψώνια, να να ζήσει. Στην περιοχή μας ε, δεν υπάρχουν μεταφορές, μόνο κάποια λεωφορεία που σταματούν κάποια στιγμή, βέβαια όλο και πιο αργά, αλλά όπως και να έχει το θέμα των μεταφορών είναι πρόβλημα, το θέμα των Ιδρυμάτων επίσης είναι σημαντικό. Το να μην έχεις ε, θεσμικά όργανα και ιδρύματα κοντά σου φορείς ε, που να σε βοηθούν ε, να κάνεις μια αίτηση για δουλειά και τα λοιπά είναι πρόβλημα. Ε, σε επίπεδο ασφάλειας τέλος. Ε, χρειάστηκαν πολλά χρόνια μέχρι να έχουμε το δικό μας αστυνομικό τμήμα, μια αστυνομία η οποία θα είναι εκεί για την, στην υπηρεσία του πολίτη και όχι στην υπηρεσία του Υπουργείου ή των Στατιστικών. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν της αστικοποίησης ε, και της στέγασης θα πρέπει να εξετάσουμε την ανθρώπινη διάσταση η οποία αυτή τη στιγμή είναι η προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα στη Γαλλία, γιατί στο παρελθόν η προτεραιότητα ήταν να στεγάσουμε τους ε, μετανάστες που ήρθαν στη Γαλλία για να βοηθήσουν στην οικοδόμησή της, αλλά ξεχάσαμε ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν κάποιες προσδοκίες και τώρα το 2010 στη Γαλλία έχουμε γκέτο. Ε, καλησπέρα. Θα είμαι και εγώ πολύ σύντομος. Θα ήθελα και εγώ να πω ότι μετά από τις ευρωεκλογέ του 2009 υπήρξε μεγάλο επίπεδο αποχής ε, σε αυτές τις ε, ε, περιοχές της Ευρώπης. Σχεδόν 80% ήταν η αποχή. Άρα σε επίπεδο δημοκρατικό είχαμε ένα έλλειμμα το οποίο το είδαμε και στις περιφερειακές εκλογές. Μία απόρριψη της πολιτικής, μία παρόλα τα χρήματα που δίνονται υποτίθεται για την ε, περιφερειακή πολιτική, ε, ο κόσμος δεν βλέπει τι ε, αποτέλεσμα έχει η Ευρώπη. Εκεί, σε αυτές τις περιοχές, είναι ένα, βρίσκεται ένα εργαστήριο, ένα φυτόριο για ανισότητες σε χώρες όπως η Γαλλία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν κανείς αν θέλει να δουλέψει ή να φοιτήσει σε ένα σχολείο κάπου, σε ένα πανεπιστήμιο ή ε, να έχει κάποια πολιτιστική δραστηριότητα πρέπει να πάει στο Παρίσι που είναι μια μισή ώρα. Έτσι λοιπόν μπορεί η περιοφέρεια αυτή να είναι η πιο πλούσια της ε, Ευρώπης, όμως ε, υπάρχουν πραγματικοί θύλακοι σε αυτή την περιφέρεια, περιοχές που δεν εκμεταλλεύονται τον τις ευκαιρίες ε, που δίνει η πόλη, η περιφέρεια, η Ευρώπη. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτεί τις ε, υπηρεσίες νεότητας, όμως ε, παρόλα αυτά είναι πολύ πολύπλοκε οι διαδικασίες ακόμα για τις ενώσει, π.χ. αθλητικού φορείς και τα λοιπά, που θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτή τη χρηματοδότηση. Είναι πολύ δύσκολο να καταθέσουν ένα φάκελο για να επωφεληθούν αυτών των χρηματοδοτήσεων. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που μας δεχτήκατε εδώ. Γνωρίζουμε ότι είστε στην υπηρεσία όλης της Ευρώπης, ότι η δική σας Επιτροπή έχει βοηθήσει σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα τις ανατολικές χώρες, ε, να ε, αναπτυχθούν οι περιφέρειες, όμως δυστυχώς στη Δύση, σε χώρες όπως η Γαλλία, υπάρχουν ακόμα πόλεις που έχουν ανάγκη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η πρόταση που έκαναν οι φίλοι μου να οργανώσουμε ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Προαστίων όπου θα έχουμε εκπροσώπους από τις διάφορες πόλεις και χώρες για να συζητήσουμε και να συγκρίνουμε τις διάφορες δυσκολίες που έχουμε κοινέ. Θα ήταν πραγματικά ευτύχημα να συμβεί. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για την υποδοχή σας και ελπίζω ότι στις δημοσιονομικές ε, στον δημο... προοπτικές σας ε, για το μέλλον ίσως θα πρέπει να σκεφτούτε όλα αυτά τα πράγματα και με βάση τη δική μας συνοικία να έχετε μια άποψη για όλες τις συνοικίες ε, σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, η κυρία Κωνσταντζα Κρέλ. Ευχαριστώ. Να ζητήσω συγγνώμη που δεν είμαστε εδώ πολύ εκ μέρους των συναδέλφων, γιατί υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση στην έναρξη αυτή της συνεδρία. Ε, χαίρομαι όμως που έχουμε λάβει αυτές τις πληροφορίες μέσω ημών. Να πω έτσι, να μετρέπει ότι αυτές οι πληροφορίες για μένα δεν είναι, για μας δεν είναι καινούριες. Ε, δεν είναι το πρόβλημα αυτό μόνο πρόβλημα του Παρισιού και των γειτονιών του είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει σε όλες τις μεγάλες πόλες. Σε κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τουλάχιστον ε, υπάρχει αυτό το πρόβλημα της ενσωμάτωσης των ομάδων πληθυσμού που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Έχουμε προσπαθήσει να βρούμε κάποιο τρόπο, κάποιο σύστημα μέσα από την ε, πολιτική συνοχή να λύσουμε αυτό το θέμα και ακριβώς ε, να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δυσκολίες. Η ενσωμάτωση νέων ε, ανθρώπων στην αγορά εργασίας, η βελτίωση της εκπαίδευσης, η δυνατότητα οι ενώσει και οι σύνδεσμοι και οι σύλλογοι να συνεργαστούν με τις ευρωπαϊκές δομές είναι πράγματα που είδαμε στο Παρίσι, τα είδε η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Μάθαμε και θετικά πράγματα. Υπάρχει στη Γαλλία η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί αυτό το σύστημα εργαλείων και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να μην να σας προτρέψω να μην σταματήσετε τις προσπάθειες. Αξίζει τον κόπο και οι άνθρωποι που τους αφορά το θέμα αυτό ε, αξίζει να τύχουν αποτελεσμάτων των προσπαθειών σας. Θέλουμε αυτό το σύστημα εργαλείων. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση να γίνεται ε, σε συνεργασία με όλους αυτούς τους ανθρώπους που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνο από λίγους. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι σημαντικό ε, να επιστήσουμε την προσοχή στο γεγονός ότι τώρα μπήκε στο, η συζήτηση το θέμα της ειφόρου ε, ανάπτυξης και της ενσωμάτωσης των, ε, ε, των πόλεων και ότι τώρα μέσα από την πολιτική συνοχή θα υπάρχει ένας προϋπολογισμός που θα καθιστά δυνατή την πρόθεση αυτών των προτεραιοτήτων. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει εντατική εργασία και συνεργασία ε, με εμά ε, και με τους ενώσεις και τους οργανισμούς ε, θα είναι καλό να είμαστε σε επαφή έτσι ώστε να έχουμε επαφή με τη βάση, να έχουμε πραγματικές εμπειρίες και γι' αυτό παρακαλώ συνεχίστε να προσπαθείτε και παρακαλώ όχι με τη βία. Είναι το πιο δύσκολο μέσο που κανείς πρέπει να χρησιμοποιεί δυστυχώς πάντοτε βλέπω σε ταινίες, στην τηλεόραση κτλ. Ε, σκηνές από, ζωές, από τη ζωή στο Παρίσι και σε, ε, στις γειτονιές του που θα μπορούσαν να ήταν καλύτερες συνθήκες αν ε, είχαμε τη βοήθεια των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Επιτρέψτε μου να πω και εγώ δύο λόγια. Επισκέπτεστε τώρα μια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ασχολείται με την περιφερειακή και την αστική ανάπτυξη. Νομίζω ότι όλα όσα είπε, ε, Κωνσταντσα, ε, σωστά είπε, όλα αυτά που λέτε μα είναι γνωστά αλλά και μα ανησυχούν ε, τα μάλα. Έτσι λοιπόν, χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήρθατε και μπορούσαμε να ακούσουμε και από σας άμεσα αυτές τις πληροφορίες από πρωτοχέρι. Τώρα συζητάμε εδώ την μελλοντική πολιτική συνοχής και τη μελλοντική ε, αστική πτυχή της πολιτικής συνοχής και όλα τα προβλήματα που σχετίζονται με την αστική ανάπτυξη και έχουν να κάνουν ε, με το κοινωνικό αποκλεισμό και τη στέρηση και όλα αυτά τα προβλήματα που απαιτούν λύσεις ε, πρέπει να ληφθούν ε, σοβαρά και στη μελλοντική πολιτική, στην ε, αστική διάστηση της πολιτικής συνοχής. Αύριο έχουμε και μία κρόση εμπειρογνωμόνων, αλλά θα και με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συζητήσουμε την κατάσταση στις ευρωπαϊκές πόλεις, θα συζητήσουμε τις προκλήσεις που τίθενται και φυσικά θα τους διαβιβάσουμε και όλα όσα μας είπατε. Επίσης, ε, το Δεκέμβριο, ο Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής ε, θα ε, έρθει εδώ να συζητήσει μαζί μας το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Έτσι λοιπόν, σας ευχαριστούμε για όλες τις πληροφορίες που προσθέσατε, όσα γνωρίζαμε ήδη από την επίσκεψή μας στη Γαλλία. αλλά μπορούμε να πούμε ότι τώρα έχουμε και άμεση ενημέρωση από όλους ε, όσους ε, υφίστανται όλα αυτά τα προβλήματα. Αλλά θέλω να σας διαβεβαιώσω στη συζήτηση ε, και στη μελλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής ε, θα δοθεί η πολύ μεγάλη εστίαση στο τι μπορεί να γίνει τοπικά στις ε, αστικές περιοχές προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλες αυτές οι προκλήσεις και τα προβλήματα που μας καταθέσατε εδώ. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όχι μόνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γι' αυτό αυτή η ανταλλαγή απόψεων μαζί σας ε, για μας ε, είναι ένα πρόσθετο επιχείρημα υπέρ του να ασκήσουμε πίεση υπέρ μιας πολιτικής συνοχής που θα απαντήσει σε όλα αυτά τα προβλήματα. Κυρίως ε, στις αστικές περιοχές αλλά και στα προάστα, στα μπανιέ. Και και θα συζητήσουμε και με τον πρόεδρο της Γαλλίας τις επόμενες μέρες. Θα του διαβιβάσουμε όλα αυτά που ακούσαμε, αλλά το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα τοπικά. Και εγώ θέλω να σας ενθαρρύνω ως συλλογή να είστε πάρα πολύ ενεργοί ε, σε σχέση με την τοπική δράση, γιατί πάρα πολλά εξαρτώνται και από εσάς. και πρέπει και εσείς οι ίδιοι να είστε ενθουσιώδεις και να αναλαμβάνετε δράσεις για να αλλάξετε την κατάσταση. Πάρα πολλά μπορούν να επιτευχθούν αν ε, υπάρχει μια τοπική κοινότητα η οποία πραγματικά θέλει να σημειώσει πρόοδο και με λίγη βοήθεια μπορείτε να κάνετε πολλά, αλλά αν ε, και εσείς ε, στρέψετε στην πλάτη σας αυτό που μπορούμε γενικά να σας προσφέρουμε από την Ευρώπη, το ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολη η κατάσταση. Έτσι λοιπόν να είμαστε σε επαφή ε, και σας απευθύνουμε και μια έκκληση να παραμείνετε και σε ενεργοί σε τοπικό επίπεδο και εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας και στη μελλοντική πολιτική να έχουμε και μέσα και δράσει που θα σας επιτρέψουν να αλλάξει η πραγματικότητα στην οποία ζείτε. Uh, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια προσπάθεια πανευρωπαϊκή ε, που υλοποιείται τώρα, αλλά και εσείς, η κοινωνία των πολιτών και οι τοπικές αρχές ε, πρέπει ε, να αναλάβετε κάποιες δράσεις, αλλά και σε εθνικό επίπεδο πρέπει να γίνουν κάποιες δράσεις, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι είναι σημαντικό όλοι μαζί να συνεργαστούμε και πάλι σας ευχαριστώ πολύ που ήλθατε εδώ και φυσικά θα σας κουβαλάμε μαζί μας, ε, στην καρδιά μας και στο μυαλό μας. Θα θυμόμαστε όσα είπατε και φυσικά θα συζητήσουμε και με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα για να διασφαλίσουμε ότι στο μέλλον ότι στις ευρωπαϊκές πολιτικές θα αποτελεί αυτό υψηλή προτεραιότητα, τα προβλήματα δηλαδή που μας παρουσιάσατε. Uh, Ξέρετε ότι πολλά έχουν ήδη γίνει βέβαια. Δεν ξέρω πόσο εσείς ε, έχετε μπορέσει να υποφεληθείτε, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε με τη βοήθεια του Κοινοβουλίου σε σχέση με το τι μπορεί να γίνει για τη στέγαση και επίσης απλοποίησαμε και την πολιτική Βέβαια τελικά θα δούμε γιατί όλα αυτά εξαρτώνται και από τόσο μεγάλο θα είναι ο ευρωπαϊκός προπολογισμό. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι μόνο το 1% του ΑΕΠ όλων των κρατών μελών. Είναι πολύ μικρός λοιπόν ο προπολογισμό, αλλά δεν είναι μόνο τα χρήματα εδώ, είναι και η δική σας συμμετοχή και η συνεργασία. Νομίζω ότι όλα αυτά μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Κύριε Ντέλη, θέλετε κάτι να πείτε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας ζητήσω να λάβετε υπόψη σας τον, χαρακτήρα έκτακτης ανάγκης. Γιατί εδώ έχουμε πολλά θέματα και πρέπει να ενεργοποιήσουμε αυτά τα ευρωπαϊκά ταμεία που θα απευθύνονται σε εσάς έτσι ώστε να μπορείτε να πραγματοποιήσετε τα προγράμματα και τα σχέδια που έχετε. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ευθύνη μας να ενσωματώσουμε αυτές τις προτεραιότητες στη μελλοντική ατζέντα. Όπως είπε και ο Ευρωπαίος Επίτροπος, αυτά τα θέματα πρέπει να τα δούμε από τον Ιανουάριο και θα πρέπει να συνεργαστούμε θα ξεκινήσουμε και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε έτσι ώστε η πολιτική συνοχής να ε, είναι κάτι από το οποίο θα αποφελούνται όλοι. Έτσι ώστε μέσα σε αυτή τη χρονιά ε, καταπολέμησης της φτώχειας να καταργηθούν αυτές οι ανισότητες. Θα προχωρήσουμε λοιπόν με έναν ενεργό τρόπο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Αντέλη. Θα ήθελα Επίσης, να σας ζητήσω να μας αφήσετε αυτά που τα έγγραφα που έχετε ε, γραπτός. Ε, θέλετε όμως το λόγο, παρακαλώ. Καλημέρα. Είμαι ο Φαρίντ Μπεραής. Είμαι πρόεδρος μιας ε, οργάνωσης ε, του kickboxing και είμαι και προπονητής. Είμαι λοιπόν από τον τομέα του αθλητισμού άκουσα όσα αυτά που είπατε, όλα όσα είπατε. Και τώρα γνωρίζουμε καλύτερα τι συμβαίνει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, έχουμε και εμείς ερωτήσεις πώς πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα από τη δική μας πλευρά μας. Έχουμε μία οργάνωση η οποία διέπεται από τον νόμο του 1901 για τις οργανώσεις και υπάρχουν διαφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη λειτουργία των οργανώσεων. Κάτι που δεν συζητήσαμε είναι ο εθελοντισμός. Είμαι προπονητής, όπως είπα, και ε, κάνουμε θελοντικά αυτή την εργασία εδώ και αρκετά χρόνια. Ε, με τους δήμους, τις περιφέρειες, τα διαμερίσματα προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε κάποιες ε, ενισχύσεις έτσι ώστε να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. και αυτό αφορά τα, τα σχολεία αλλά και τους νέους που βρίσκονται ήδη στην αγορά εργασίας και προσπαθούμε πάντα να είμαστε παρόντες ε, τόπου Και αυτό συνέβη και το 2005. Και δεν τα παρατάμε ποτέ. Ε, βλέπουμε ότι τα πράγματα γίνονται όλο ένα και πιο δύσκολα, όμως είμαστε υπομονητικοί. Όμως ε, φτάνει κάποια στιγμή που χάνουμε αυτή την ανέργεια που έχουμε και αυτό συμβαίνει πιστεύω ε, στην νεολαία σε όλη την Ευρώπη. Εμείς προσπαθ, πλαισιώνουμε την νεολαία που έχει όρεξη για δραστηριότητες εξωσχολικές, να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, όμως είναι πολύ δύσκολο για εμάς να μπορούμε να χειριστούμε όλη αυτή την ενέργεια της νεολαίας. Ε, σας ευχαριστώ και πάλι που μας δεχτήκατε εδώ σήμερα. Μπορούμε να έχουμε κοινά προγράμματα, κοινά σχέδια. Θα προσπαθούμε να έχουμε κοινά σχέδια με άλλες οργανώσεις άλλων χωρών όπως το Βέλγιο, η Γερμανία κτλ. Προσπαθούμε επίσης να εναρμονίσουμε τον αθλητισμό έτσι ώστε να υπάρχει παντού σε όλες τις χώρες η ίδια λειτουργία. Όμως ε, η έννοια του εθελοντισμού δεν υπάρχει παντού. Είναι κάτι με ιδιαίτερα τοπικό χαρακτήρα. Θα θέλαμε κάποιες απαντήσεις, έστω και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε να μπορέσω να γυρίσω στο κλεισί Σουμπουά και να πω στους ε, μαθητές μου ότι η Ευρώπη θα τους στηρίξει, θα τους βοηθήσει και θα είναι παρούσα. Νομίζω έτσι θα κάναμε ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Και θα είναι μια ε, κατάσταση από την οποία θα υποφεληθούν όλοι. Δεν προσπαθώ εδώ να σας πουλήσω κάτι, όμως νομίζω ότι θα κερδίσουμε πολλά από αυτό. Πρέπει όμως να σας πω ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή μέσα σε αυτό το, το, τον κόσμο και σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Σας ευχαριστώ. Θα συνοψίσω σύντομα, γιατί πρέπει να κλείσουμε και τη συνεδρίαση. Φυσικά γίνονται πολλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως, πολλά πρέπει να γίνουν και σε τοπικό επίπεδο. Θα δείτε τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στον επόμενο χρόνο για τους νέους και αυτό σχετίζεται με την στρατηγική που έχει στην ατζέντα και που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που στήριξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη. Μία ε, πρωτοβουλία σημαία είναι οι νέοι άνθρωποι. Έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη υποστήριξη από το ευρωπαϊκό επίπεδο προς τους νέους και προς τη νέα γενιά. Επίσης, στον προπολογισμό για την επόμενη χρονιά δεν έχει ληφθεί ακόμα η τελική απόφαση, όμως υπάρχουν προγράμματα για τους νέους ανθρώπους και βρίσκονται πολύ ψηλά στην ε, ατζέντα. Τούτου λεχθέντος, θα ήθελα να σας θαρρύνω μέσω των ε, βουλευτών σας ε, να διατυπώσετε τις ερωτήσεις σας έτσι ώστε να λάβετε πληροφορίες για να δείτε ποια είναι τα ευρωπαϊκά προγράμματα και σχέδια που υπάρχουν Υπάρχουν πολλά για τον αθλητισμό, για τις άλλες δραστηριότητες και θα μπορούσατε ίσως να ε, υποφεληθείτε από αυτά ε, και ίσως δεν ξέρετε πώς. Ε, μπορούμε να σας δείξουμε λοιπόν ποιος είναι ο τρόπος και επίσης μπορείτε να μας πείτε ποιες είναι οι προσδοκία σας και να βρείτε διάφορες πληροφορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να δείτε τι κάνει λοιπόν η Ευρώπη για τους νέους αυτό που είναι σαφές είναι ότι οι νέοι στα επόμενα χρόνια θα είναι στο κέντρο της εστίασης του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλείνοντας λοιπόν, θα ήθελα να σας πω να κρατήσουμε την επαφή και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Η κυρία Δέλη θέλει το λόγο. Για να συμπληρώσω κύριε Πρόεδρε. Το επόμενο έτος είναι το έτος εθελοντισμού. Ευρωπαϊκό Εθελοντισμού ίσως λοιπόν είναι μια ευκαιρία να αξιοποιήσετε τις εμπειρίες σας ε, και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα συναντηθούμε και θα συζητήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε βάσει και του προπολογισμού για να απελευθερώσουμε το τάδι το δίνα πρόγραμμα. I would like to, to close the θα ήθελα τώρα εδώ να κλείσω τη συνεδρίαση και πάλι θέλω να σας ευχαριστήσω. Ακόμη και αν είμαστε πολύ λίγοι όσοι απομείναμε, καταλαβαίνετε ότι ε, σας σκεφτόμαστε, θα είμαστε σε επαφή και καλή επιστροφή.